για τις ψηφοφορίες που μόλις ολοκληρώσαμε. Καταρχάς, ε, επεξηγήσεις ψήφου για την ψηφοφορία για την έκθεση του Chris Davis ε, για την ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπόδων ανθρακούχων εκπομπών μέχρι το 2050. Ο πρώτος ομιλητής, ο κύριος Καμίνσκι, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι στόχοι που επισημαίνονται στην έκθεση είναι σαφώς ε, στόχοι που είναι αρκετά γενναιόδοροι. Η περιβαλλοντική προστασία είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί όλους και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφάτως δείχνει να επιβάλλει πάρα πολύ ευστηρά ε, λύσεις υπέρ του περιβάλλοντος ε, σε τομείς τους οποίους ε, δεν είναι κοινοί οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες που ρηπαίνουν πολύ περισσότερο, όπως για παράδειγμα η Ινδία και η Κίνα. Δεν θα πρέπει δεν ε, να βλέπουμε και το γεγονός ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το τίμημα για όλους αυτούς τους ευσεβείς πόθους και τους ευγενείς σκοπούς που αναλαμβάνουμε θα το πληρώσουν οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Συνεπώς, ε, παρά το γεγονός ότι συμφωνώ με τα επιχειρήματα δεν μπόρεσα να υπερψηφίσω. Ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Φραντσέσκο Ντεαντζέλης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έγκριση του συγκεκριμένου κειμένου θα πρέπει να συνεισφέρει να αυξηθεί το επίπεδο των επενδύσεων και να διασφαλίσουμε έτσι και το βιομηχανικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να δώσουμε στο βιομηχανικό τομέα τα απαραίτητα κίνητρα προκειμένου να προάγουν επενδύσεις οι οποίες μπορούν να ευνοήσουν την οικονομική ανάπτυξη και μπορούν ταυτόχρονα να μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Μία οικονομία χαμηλών εκπομπών ε, άνθρακα σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μειώσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε άλλο θα πρέπει να την ενισχύσει θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις απαραίτητες επενδύσεις προκειμένου να ευνοήσουμε την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ε, ενέργειας για να έχουμε αποταμίευση και καθαρή ενέργεια. Η Ευρώπη θα πρέπει να επιταχύνει σε αυτό το τομέα αν δεν θέλει να μείνει ε, πίσω. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια πραγματική πράσινη οικονομία η οποία μπορεί να δημιουργήσει ανάπτυξη και βιώσιμη ανάπτυξη εν γέννη. Ευχαριστώ κύριο Σόνικ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την έκθεση Davis, σε σχέση με τις ε, χαμηλές ε, εκπομπές άνθρακα, ανταγωνιστική οικονομία λοιπόν ε, μέχρι το 2050, θα πρέπει να δούμε πρώτον το κόστος της μείωσης και η ανασφάλεια που θα προκληθεί στη βιομηχανία είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί πρέπει να τους δώσουμε ένα σαφές μήνυμα. Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν συμφωνίε πολλών ετών ε, για τι εκπομπέ του άνθρακα, τι οποίε τώρα τροποποιούμε. Όμω η βιομηχανία είχε κάνει τι επενδύσει τη με αυτόν τον ορίζοντα, τον ορίζοντα του 2020. Αυτή λοιπόν η ρυθμιστική ασφάλεια σε ό,τι αφορά την, ε, τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα υπάρχει περίπτωση να χαθεί. Ο κύριος Μπίλαν τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ψήφισα κατά της έκθεσης. Κατά της στρατηγικής αυτής, διότι πραγματικά θα έχετε τα αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα. Ούτε και η πολωνική κυβέρνηση ενέκρινε την ε, συμφωνία αυτή, γιατί θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν το νωρίτερο τρία ε, χρόνια μετά τις ε, διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Δεν γνωρίζουμε όμως ποια θα είναι η εικόνα της οικονομίας ευρωπαϊκής της επόμενες δεκαετίες. Η αφαίρεση του άνθρακα από την βιομηχανία θα πλήξει την πολωνική οικονομία που βασίζεται ε, στις άδειες εμπορίες εκπομπών. Και θα μειωθεί και το βιωτικό επίπεδο, το επίπεδο διαβίωσης του μέσου Πολωνίου ως αποτέλεσμα αυτής της νέας νομοθεσίας. Γι' αυτό λοιπόν διαφωνώ με τις ε, αρχές της ε, Κομισιόν σε ό,τι αφορά και τις ευρωβουλικές εκπομπές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η μείωση ε, των ε, ε, αερίων θερμοκηπίου είναι ένας βασικός στόχος της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε λανθασμένα κίνητρα. Πρέπει καλύτερα να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το καλό των φυσικών μας πόρων χρόνο να μην μειώνουμε ε, και να μην αποκλείουμε ορισμένους τομείς διότι υπάρχουν αποτελέσματα που δεν αποδεικνύονται επιστημονικά και κατά τη γνώμη μου η γεωργία δεν είναι πρόβλημα του προβλήματος αλλά της λύσεως γιατί και εκεί υπάρχουν διοργασίες μεταλλαγής ε, ορισμένων αερίων οπότε θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις απόψεις Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπασέσκου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση διότι υποστηρίζω τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συνεχίσουμε τις ε, διεθνείς ε, ε, συμβάσεις για την αλλαγή του κλίματος. Θεωρώ ότι η Ευρώπη πρέπει ε, να προσαρμοστεί με βάση και τους στόχους της Ευρώπης 2020. Έτσι θα έχουμε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και μια ε, σοβαρή οικονομική στρατηγική. Η χώρα μου υποστηρίζει τα θέματα αυτά, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ρουμανία και άλλε χώρε τη Ανατολική Ευρώπη θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει το ορόσημο του 1999 για, τις μελλοντικές, για τα μελλοντικά πλαίσια, έτσι ώστε να έχουμε μία εικόνα του τι ακριβώ έχουν επιτύχει τα κράτη-μέλη αυτά για τη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Επίση, θεωρώ ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε το πρόγραμμα για την μεταφορά των πλεονασμάτων από το ε, σύστημα του Κιώτο και επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να πείσουμε για μεγαλύτερη συνένεση από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Ο κύριος Σονκέλη στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, πολλές καλές συστάσεις ε, περιέχει η έκθεση, αλλά και επίμαχες συστάσεις μεταξύ άλλων. Τελικά, καταφέραμε να φτάσουμε σε μια ικανοποιητική ε, έκθεση. Επειδή βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αν θέλουμε να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή οικονομία χρειαζόμαστε νέες θέσεις εργασία, νέε βιομηχανίε, Ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και απ' την άλλη βέβαια έχουμε και τι ανησυχίε μα για το περιβάλλον. Πρέπει να βρούμε σωστή ισορροπία. κάποιε προτάσει ενδέχεται να βλάψουν την οικονομία και ίσω απορρίφθηκαν κάποιοι που δεν θα έβλαπαν την οικονομία. Το στόχο, ο στόχο είναι πάντω ε, ε, να δούμε τι θα κάνουμε απέναντι σε άλλε χώρε, κυρίω όπω είναι η Κίνα και η Ινδίνα. Και θα πρέπει, πιστεύω, παγκόσμια να δρώσουμε συνολικά για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Αυτή είναι η πρόκληση. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίο ομιλητή είναι ο κύριο Τάνοκ. Και εγώ, όπως και η ομάδα μου, ε, απήχαμε σε σχέση με την έκθεση αυτή η ιδέα ε, της έκθεσης είναι καλή για την καταπολέμηση αλλαγής του κλίματος ε, και για την ε, εξοικονόμηση υδρόγων ανθράκων. Όμως ζητάει η έκθεση από την Κομισιό να προτείνει μέτρα για την επίτευξη των στόχων του 2030 πάρα πολύ γρήγορα και επίσης ζητάει από την Κομισιό να κάνει πιο ριζικές και παρεμβάσει για να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίε του συστήματο εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών. Παραδείγματο χάρη, ε, κάποιες ε, άδειε και στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών πρέπει να συμπεριληφθούν. Τελικά έχει μετριαστεί, ε, έχει κάπως αποδυναμωθεί η πρόταση. Το συμβαστικό πακέτο εμεί θεωρούσαμε ότι ήταν πιο αποτεκτό αλλά τελικά σαν ομάδα δεν νομίζουμε ότι μπορούμε να δεχθούμε τις βασικές διατάξεις τη έκθεση στον τομέα της γεωργίας και της περιφερειακής χρηματοδότησης εξού και απήχαμε. Σας ευχαριστώ. Τώρα περνάμε σε επεξηγήσεις ψήφου για του ιστοτόπους που υποκινούν διακρίσεις και κυβερνητικέ αντιδράσεις. Κύριε Καμίνσκι, για το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Αυτό το οποίο πρόσφατα συνέβη στην ε, Ολλανδία με ένα πολιτικό κόμμα το οποίο υποστηρίζει και την ε, κυβέρνηση της χώρας έχει να κάνει με την ε, υποκίνηση μίσους ε, κατά των ε, μειονοτήτων στην χώρα αυτή για πολιτικό όφελος. Χαίρομαι που βλέπω ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ολλανδία ξεσήκωσαν την αντίδραση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε αυτά τα κρούσματα μόνο στην Ολλανδία φωνές κατά Πολωνών μεταναστών ε, ακούγονται και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και μάλιστα κάποιοι από τους εκπροσώπους ε, κομμάτων εδώ στο Κοινοβούλιο έχουν εκφράσει αντίστοιχες ιδέες. Πρέπει να πάψει αυτή η αντιπολωνική ρητορική. Ο κύριος Στάνιελ Χάναν για να Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε το σώμα είναι, έχει μια αιμονή με τις ψήφους για το κλίμα. Έχουμε ένα σωρό ψηφίσματα και εκθέσεις που θέλουν να δείξουν ότι ε, είμαστε σοβαροί και ψηφίζουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν επιπτώσει στον πραγματικό κόσμο. Όσο μεγαλύτερο γίνεται η οικονομική κτήση, όσο περισσότερο ασχολούμαστε με όλα αυτά τα θέματα. Η Ελλάδα καταραίει και εμείς ε, καθόμαστε και ασχολούμαστε για, με μια ιστοσελίδα για τις κάτω χώρες και δεν ξέρουμε ούτε ποιοι είναι οι γράφαντες αυτές τις ιστοσελίδες. Τους δώσαμε διαφήμιση ε, που ούτε το φανταζόντουσαν. Δεν καταδικάζουμε ούτε καν ε, το κόμμα ε, που έχει υποκινήσει όλα αυτά. Δεν καταδικάζουμε το κόμμα του Ολλανδού Πρωθυπουργού. Ε, φαντάζομαι ότι θα σπαταλήσει πολύ χρόνο και θα αρχίσει να εξηγεί στους υπολείπους τι γίνεται και μετά θα τους πει ότι κοιτάξτε να δείτε έχω και μια χώρα να διοικήσω ο ένας καταδικάζεται και μετά κάποιος άλλος πρέπει να παρουσιάσει ένα ψήφισμα θα ήμασταν πολύ πιο σοβαροί εάν, και αξιόπιστοι εάν σταματήσουμε να χαϊδεύουμε ένα στα αυτιά του άλλου και να ασχολούμαστε συνέχεια με τέτοια θέματα τα οποία ε, είναι ασήμαντα στην πράξη και να ασχολούμαστε με ψηφίσματα που ενδιαφέρουν τον πραγματικό κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσαμπασόκα. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση αυτή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μια χώρα η οποία έχει ένα, μια ισχυρή δημοκρατική και φιλελεύθερη παράδοση. Αναφέρομαι στις κάτω χώρες, διότι ε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα καθαρά ρατσιστικό ιστότοπο ε, με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης που υποκινεί μίσος μεταξύ πολιτών των άλλων κρατών μελών. Ε, είναι δεκαστέα φυσικά αυτή η πρακτική, ακόμα και αν πρόκειται για πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά επειδή ακριβώς ο στόχος είναι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώ ότι κάτι πρέπει να γίνει για αυτό το λόγο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τις διαιρέσεις. Ε, δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι οι καλοί και οι κακοί πολίτες, διότι ε, όπως έχουν οι συνθήκες χρειαζόμαστε περισσότερη αλληλεγγύη και περισσότερη Ευρώπη και δεν θα πρέπει να υποκινούμε το μίσος. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ πολύ. Το ψήφισμα αυτό είναι ένα ψήφισμα το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη ε, μιας διαδικασίας. Είναι το ψήφισμα ε, που ξεκινά κυρώσεις ε, για ε, ξενοφοβικές ιστοσελίδες ε, και για υποκίνηση μίσου. Είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνουμε κάτι τέτοιο και θεωρώ ότι είναι πονίδιστο το γεγονός. Αναφερόμαστε σε μια κυβέρνηση συνασπισμού, έχουμε φιλελευθέρους και χριστιανοδημοκράτες που συμμετέχουν σε αυτή την κυβέρνηση και η κυβέρνηση δείχνει ανοχή προ αυτή τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν θα ήθελα να γίνει ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο θα δημιουργήσει ανταγωνισμό μεταξύ πολιτικών ομάδων, αλλά υπάρχει ευθύνη από τους χριστιανοδημοκράτες και τους φιλελευθέρους και θα πρέπει να την αναλάβουν. Θεωρώ ότι μέσω της αγωγής του πολίτη, μέσω μιας κατάλληλης εκστρατεία περιορισμού του φαινομένου θα μπορούσαμε ίσως να ε, το πατάξουμε, διότι δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, ειδικά σε καιρούς κρίσης, διότι η κρίση μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα με τα δημοκρατικά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό τώρα η κυρία Ρόιτοβα. Ευχαριστώ.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 ε, υπάρχει ε, μία κατα... Ε, παραβίαση της δημοκρατίας και θα βλέπουμε ότι υπάρχει μία επίθεση κατά όλων των Ευρωπαίων γι' αυτό και σήμερα δεν πρέπει να αποδεχθούμε το ψήφισμα αυτό αλλά να συνεχίσουμε να πιέζουμε τον Πρωθυπουργό της Ολλανδίας διότι αυτό το είδος της ε, διάκρισης δεν είναι επιτρεπτό και είναι αντίθετο με τις ελευθερίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση δεν έχει δείξει ε, σαφή επιχειρήματα και η Ολλανδία χρησιμοποίησε την ε, κατάσταση στην Ευρώπη για να αγοράσει ε, ε, εξοχικές κατοικίες στην Τσεχία οπότε θα θέλαμε η κοινωνία των Ολλανδίας να τεθεί κατά αυτής της ξενόφοβης πολιτικής. Ο επόμενος τον κύριο Στάντλερ. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα καταψήφισα αυτό το ψήφισμα διότι είμαι της ε, γνώμης ότι κάθε Ευρωπαίος πολίτης έχει το δικαίωμα ε, να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα υποβάλει το παράφωνο ή την προσφυγή του και αυτό έχουμε διαπιστώσει και στο παρελθόν. Μπορεί να γίνει μέσω της εφημερίδας. Δεν είναι θέμα ε, πολιτικού σαβουάρ και εδώ απευθύνουμε στον κύριο Καμίνσκι. Δεν είναι σωστό να αναφέρεται κανείς σε ε, κράτη είτε είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είτε εκτός αυτής. Ιδίως για την ε, Πολωνία διότι οι δικές μου εμπειρίες με την Πολωνία είναι τελείως διαφορετικές η εγκληματικότητα δεν είναι εθνική, είναι διεθνής Ευχαριστώ πολύ. Ο Σαλβατόρη Ιακολίνο τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σαφώς και είναι χρήσιμη μια πρόταση κοινού ψηφίσματος για ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα της διάκρισης κατά των ανθρώπων που κανονικά θα έπρεπε να ενταχθούν και να τους καλοδεχτούμε εκεί ε, όπου υπάρχει δυνατότητα να βρουν μια θέση εργασίας και να μπορέσει να υπάρξει ίσως και πανένωση των οικογενειών τους. Η ευρωπαϊκή υπηκότητα είναι ένα θέμα μεγάλης αξίας και θα πρέπει σαφώς να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Θα πρέπει να ε, ξαναδώσουμε όθηση στο θέμα της υποδοχής και της ένταξης. Υπάρχουν οδηγίες όπως για παράδειγμα η 32 του 2004 που είναι ουσιαστική σημασία για το ζήτημα και όταν εμείς προετοιμαζόμαστε το 2013 να εορτάσουμε το Ευρωπαϊκό Έτος για τους πολίτες, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι θα πρέπει να άρουμε και οποιοδήποτε εμπόδιο αποτελεί πρόσκομα προς όλη αυτή τη διαδικασία. Το διαδίκτυο είναι ένα βασικό μέσο γνώσης και πληροφόρησης, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις και απαιτήσει που θα πρέπει να τηρούνται από αυτούς που το χρησιμοποιούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια, κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έπρεπε να πάρω το λόγο γιατί η διάσκεψη των Πρόεδρων αποφάσισε ότι μόνο οι επικεφαλείς πολιτικών ομάδων θα μπορούν να, να λάβουν το λόγο στη διάρκεια της συζήτησης. Αυτό σήμαινε ότι δεν είχαν πλέον ελευθερία έκφρασης οι υπόλοιποι βουλευτές. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο να μας βάζουν τέτοιες ταμπέλες αρνητικά στερεότυπα οδήγησαν ε, στο ολοκαύτωμα, στη σφαγή της Ρεμπρένιτσα. Είδαμε τη σφαγή επίσης στην Ορβηγία πέρυσι το καλοκαίρι και πραγματικά οι εκπρόσωποι, ε, μάλλον αυτό το Ολλανδικό Κόμμα εκπρόσωποι το οποίο βρίσκονται εδώ δεν έχουν αποστασιοποιηθεί από την ε, στάση του ΠΒΒ. Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε τις ακρότητες, τους εξτρεμισμούς, την ξενοφοβία. Και η Ολλανδική κυβέρνηση έχει κάνει κι άλλα. Παραδείγματο χάρη έχει μπλοκάρει την είσοδο τη Ρουμανία ε, στην προσχώρησή τη ε, στο Σέγγεν και την πρόσβαση στην αγορά εργασία. Επόμενο ομιλητή, ε, Μπίλαν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με την θέση της Επιτρόπου Ρέντινγκ Η καταγγελία σε βάρος εργαζομένων από τρίτες χώρες όπως την Πολωνία παραβιάζει ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πρωτοβουλία αυτή δείχνει ακραία ε, ξενοφοβία και μυσαλλοδοξία. Και είμαι αντίθετος. Έχουμε ανησυχητικά φαινόμενα. Βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα από την ε, Ολλανδία. Μια χώρα όμως που είχε καλές σχέσεις με την Πολωνία για πολλά χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που μας έχουν βοηθήσει και όλους όσους λένε ότι οι Πολωνοί μετανάστες πάντα είναι, ε, έχουν τις καλύτερες δυνατές προθέσεις. Ελπίζω να μην έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα σε οποιαδήποτε άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρέπο τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, είμαι υπέρ αυτής της ε, πρότασης ψηφίσματος διότι θα πρέπει το Κοινοβούλιο να είναι απερίφραστο στην καταδίκη οποιασδήποτε ε, διακριτικής ε, μεταχείρισης. Δεν θα πρέπει ε, να επιτρέπουμε τέτοια φαινόμενα. Μιλάμε για ανοιχτή υποκίνηση σε μίσος και για διακριτική μεταχείριση αυτήν στο σελίδα του ΠΒΒ. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτό, γιατί αντίστοιχε δραστηριότητε ενδέχεται να εξαπλωθούν και σε άλλε χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να οξύνουμε τι προκαταλήψει ε, να έχουμε την καλή Δύση και την κακή Ανατολή βάσει εθνικών ε, διακρίσεων, να μιλάμε για τους ε, τεμπέλιδες του Νότου και για τους εργατικούς του βόρα Πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για να πάψουν αυτά τα χάσματα και αυτή η περιχαρακώση. Ευχαριστώ πολύ. τώρα. Θα μπορούσε κανείς ε, να ε, χαρακτηρίσει σεξπυρικό το θέαμα το οποίο βλέπουμε εδώ με αυτό το site ε, της, του Ολλανδικού κόμματο. Εντάξει, δεν είναι και ό,τι πιο εγκομιαστικό και αξιέπαινο, αλλά αν ένα Ολλανδικό κόμμα, το οποίο ήταν πάντοτε αντίθετο στην νόμιμη ή στην παράνομη λαθρομετανάστευση, ιδίω από την Ανατολική Ευρώπη, αν υπάρχει ένα τέτοιο κόμμα, τότε αυτό το κόμμα έχει το δικαίωμα να κάνει κάποιες δημοσκοπήσεις ζητώντα την άποψη των ε, ψηφοφόρων του ή των πολιτών και δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει σε αυτά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί εδώ μιλάμε για την ελευθερία έκφρασης και όταν παρεμβαίνει το Κοινοβούλιο, όταν αναμειγνύει σε τέτοια θέματα αυτό ε, δίνει πολύ κακά μηνύματα και ε, δεν θα καταφέρουμε να προθέσουμε αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ κύριο Σπόσελ ο κύριος Βίλντερς ε, το κόμμα του και ο, ε, ε, η ιστοσελίδα τους είναι ακραίοι πολιτικοί και γίνονται ανεκτοί. Ενώ η ουγγαρική κυβέρνηση καταπολεμά τους εξερμιστές της δεξιάς. Ενώ η Ολλανδική κυβέρνηση στηρίζεται από αυτούς τους και πρέπει και κάποια στιγμή να γίνει ανοιχτά συζήτηση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να πω όμως ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι έχουν εκφραστεί κατά αυτή της ιστοσελίδα. Θα ήθελα όμως αυτό να γίνει συλλογικά από την Ολλανδική κυβέρνηση και δεν είναι δυνατόν να ανέχεται κανεί αυτή την κατάσταση. Ελπίζω ότι όσο ε, νούπο θα υπάρξει στην Ολλανδία μια κατάσταση που θα του είναι αντάξια ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ευχαριστώ Φίλιπ τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εάν ένας Πολωνός ή άλλος πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί αντικείμενο επίθεσης ε, δεν είναι σωστό κάτι τέτοιο. Πολλοί κόσμος είναι απλώς εργαζόμενος. Αλλά ποιος ήταν ο στόχος αυτής της ιστοσελίδα, Δεν ήταν ξενοφοβικό θέλουν να προσπαθήσουν να εντοπίσουν μια σειρά από προβλήματα. Εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι η Σέγγεν δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Η Σέγγεν με το άνοιγμα των εσωτερικών συνόρων ήταν ένα δώρο στο οργανωμένο έγκλημα. Και αντί να συμπεριφερθούμε ως ε, δικαστήριο της ε, πολιτικής ε, τάξης και να ηθικολογούμε εδώ χωρίς λόγο, θα πρέπει να σοβαρευτούμε και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών λαών. Ευχαριστώ πολύ. Επεξηγήσεις ψήφων τώρα για τα ψήφισμα για τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία. Ο κύριος Καμίνσκι έχει το λόγο πρώτος. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτό που διαπιστώσαμε στη Ρωσία δεν μπορούμε να το αποκαλούμε από τεχνική σκοπιά εκλογές. Ε, ναι, εντάξει, υπήρχαν κάλπες, υπήρχαν και κάποιοι υποψήφοι και οι ψηφοφόροι μπορούσαν να μεταβούν στα εκλογικά τμήματα για να ψηφίσουν, αλλά ακούμε ότι ακόμα και σε πολύ μεγάλες πόλεις υπήρχαν πάρα πολλές παρατυπίες. Ε, αυτό ε, δεν είναι όμως ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να μιλούμε για ελεύθερες εκλογές. Υπήρξαν υποψήφοι οι οποίοι πραγματικά απειλήθηκαν. Και ε, ο, ε, κόμματα δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στις εκλογές. Δεν μπορώ λοιπόν να υπερψηφίσω το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καταδικάζει μεν τα όσα συνέβησαν στη Ρωσία, αλλά δεν φτάνει ως εκεί που θα έπρεπε. Θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο επικριτικοί, να επικρίνουμε τους Ρώσου οι οποίοι δεν είναι δημοκρατία. Ο κύριος Χάναν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάθε χώρα νιώθει την πίεση της ε, ε, διπλωματίας, ε, της ενεργειακής διπλωματίας, της εκδίκησης, η Λευκορωσία, η Γεωργία, ε, το πιο εντυπωσιακό το 2008 και το Αζερβαϊτζάν. Και δεν χρειάζεται καν να είναι γείτονα τη Ρωσία για να το νιώσει. Εμεί είχαμε παρενόχληση του πρέσβη μα, απελάθηκαν και κάποιο διπλωματικοί υπάλληλοι του Ηνωμένου Βασιλείου. Για ποιο λόγο, τι έχει να κερδίσει το Κρεμλίνο από τέτοια συμπεριφορή. Νομίζω ότι η απάντηση ε, έγκυται σε αυτό που έλεγαν οι Γερμανοί ιστορικοί πριμάτε είναι πολιτικ. Ουσιαστικά εξάγουμε τις εσωτερικές μας αντιθέσεις. Είναι ένα καθεστώς το οποίο συνεχίζει να εφαρμόζει την τακτική του Διέρη και Βασίλευε και να δημιουργεί προβλήματα στα σύνορά της. Γι' αυτό ακριβώς και το καθεστώς στη Ρωσία ε, δεν θα έπρεπε να μας απασχολεί απλώς και μόνο ε, για να το συζητάμε, αλλά θα πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο για την εξωτερική μας πολιτική με τη Ρωσία. Ο κύριος Ουσπάσκη. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί ήμουν παρατηρητής των προεδρικών, μάλλον των εκλογών στη Ντούμα, αλλά και των προεδρικών εκλογών και είχα τη δυνατότητα να συνομιλήσω με αρκετούς υποψήφιους. Κανείς δεν εξέφρασε ενστάσεις και αντιρρήσεις. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι δεν ήταν δίκαιες οι εκλογές. Είμαι επίσης πεπισμένος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να υπαγορεύει τις απόψεις του σε άλλους. όταν έχουμε παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ε, βάζουμε χειροπέδες ε, σε ανθρώπους και τους απαγορεύουμε να συναντήσουν ε, τους ψηφοφόρους τους και όταν βλέπουμε δυσφήμιση και συκοφαντία στην τηλεόραση κατά κάποιων ανθρώπων ούτε καν συγκαλύπτονται αυτά τα εγκλήματα που διαπράττονται κατά πολιτικών αντιπάλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε χρόνο σύρονται στα δικαστήρια άνθρωποι και έχει δημιουργηθεί και ένας μηχανισμός που θα επιτρέπει ε, το να λάμψει αλήθεια μετά από 10-15 χρόνια και αφού έχει καταστραφεί η σταδιοδρομία των ανθρώπων αυτών. Στάντλερ τώρα, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερος ότι μίλησε ήδη ο κύριος Μπουσπάσκη διότι και εγώ μπορώ να επιβεβαιώσω αυτά που δήλωσε. Ήμουν παρατηρητή στη Ρωσία και τα ίδια είπε και ο συνάδελφος Νταγκαρντίνη. Ε, όποιος ε, ε, κατέκρινε την ψηφοφορία θεωρείται ότι είναι ανόητος. Οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να φέρουν την ελευθερία εκφράσεως της γνώμης στην Ρωσία δεν είναι δημοκρατική εδώ. Οι Ρώσοι ξέρουν να οργανώσουν τη δημοκρατία τους και θέλουν σταθερότητα με τις εκλογές αυτές. Δεν θέλουν να επανέλθουν στην εποχή του Γέλτσιν όπου όλα ε, υπήρχαν πάρα πολλές εισαγωγές από δυσμάς και πολλοί ολιγάρχες οι οποίοι πλούτησαν ξαδιάντροπα. Ευχαριστώ Κύριο Μπίλαν. Νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι οι δύο προηγούμενε παρεμβάσει έδειξαν πόσο αποτελεσματικά μπορεί η Ρωσία να ασκεί την επιρροή τη. Το πρόβλημα τη Ρωσία ε, σήμερα είναι ότι δεν υπάρχει φυσικά πολιτική πολυφωνία, το οποίο είναι σαφέ και φυσικά το γεγονό ότι δεν υπάρχει ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωση. Τα αποτελέσματα βεβαίω των εκλογών, επειδή δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν όλοι οι υποψήφοι, δεν μπορούν να θεωρηθούν δίκαια και τίμια το γεγονός ότι παραβιάζει ο εκλογικό νόμος είναι κάτι το οποίο χρήζει περαιτέρω ανάλυσης. Ωστόσο υπάρχει ένα μεγάλο επίτευγμα, υπάρχει μία, ε, το κίνημα αυτό στη ρωσική κοινωνία, το γεγονός ότι προσπαθούν να αποφασίσουν για την ίδια τους τη μοίρα και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει ε, να γίνει αντιληπτό από τον τρόπο με τον οποίο κυβερνά η χώρα το καθεστώ, ε, τη χώρα το καθεστώς. Θα πρέπει να ξεκινήσει διάλογος με την προδημοκρατική αντιπολίτευση και θα πρέπει να υπάρξουν και κυρώσεις για τη Ρωσία οι κανόνες για τη συμμετοχή των πολιτικών κομμάτων θα πρέπει να πλουστευθούν και οι Ξέλες θα πρέπει να θέσουν όρους για τη συνεργασία με τη Ρωσία. Ευχαριστώ. Γι' αυτό και υπερψήφισα το ψήφισμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρέπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να διαπιστώσουμε τις σημαντικές οι οποίες επετέχθηκαν εις ε, την ε, Ρωσία με από την εποχή του κομμουνισμού δεν προχώρησε η εξέλιξη διότι ε, δεν υπήρχε σοβαρός αντίπαλος για τον κύριο Πούτιν. Μετά τις εκλογές βλέπουμε ότι η κοινωνία των πολιτών έχει δραστηριοποιηθεί με την άδεια του Πούτιν. Δηλαδή πρέπει να αντιληφθούμε ότι η Ρωσία του Πούτιν δεν είναι η ίδια με προ 12 ετών όταν αυτός ε, ε, ήρθε στην αρχή. Ε, δεν θα υπάρξει βέβαια μία επανάσταση σαν την Αραβική Άνοιξη στη Ρωσία. Θα πρέπει η χώρα να εκδημοκρατιστεί μόνη της και θα πρέπει να στηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών να διατηρήσει επαφές με τη Δούμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα το ψήφισμα αυτό, λέει κύριε Αντρική, είναι παρότι δεν πιστεύω ότι αξιολογεί ορθά τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών ε, στη Ρωσία. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προβεί σε μια αξιολόγηση των εκλογών η οποία είναι ξεκάθαρη. Δεν ήταν ελεύθερες ούτε δίκαιες οι εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι οι εκλογές του Δεκεμβρίου της προηγούμενης χρονιάς ε, για τη Δούμα και οι ε, φετινές εκλογές, ε, οι προεδρικές εκλογές είναι αμφισβητήσιμες και η νομιμοποίηση των υποψηφίων και των νικητών τελικά είναι επίσης αμφισβητήσιμη. Λογικό είναι λοιπόν κάποιοι συνάδελφοι να προτείνουν ότι κάποιοι νόμοι πρέπει να αλλάξουν και αυτό πρέπει να αναφέρεται και στο ψήφισμα, μετά τι εκλογέ αυτές, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει γίνει ε, διαφορετική η Ρωσία. Εμεί θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αλλά και να δείχνουμε σεβασμό απέναντι στη χώρα αυτή. Και εμεί, οι Ευρωπαϊκοί και οι άλλοι διεθνεί οργανισμοί. Ευχαριστώ. Κριστίνα Όγιουλαν τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος και αυτό κυρίως διότι συμπεριελήφθησαν στο ψήφισμα πολλές σημαντικές τροπολογίες. Και εγώ και ο πρόεδρος της ομάδας μας, ο Γκίφερ Χόφστατ, καταθέσαμε σημαντικές τροπολογίες ζητώντας, τονίζοντας μάλλον, ότι οι προεδρικές εκλογές στη Ρωσία δεν ήταν ελεύθερες ούτε δίκαιες. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά πρέπει να καταλήξει στα συμπεράσματά της, πρέπει να αποφασίσει κατά πόσο ήταν νόμιμες οι εκλογές άρα κατά πόσο και ο εκλεγής πρόεδρος είναι νόμιμος, νομιμοποιείται από το αποτέλεσμα των εκλογών. Πριν από κάποιες ημέρες ε, διεξήχθη ακρόαση, ο κύριος Κασάνφ, ο κύριος Κασπάροφ ε, ήταν παρόντες στην ακρόαση αυτή και ορισμένοι συνάδελφοι τους έθεσαν το ερώτημα μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά να συνεχίσει να έχει σχέσεις ε, σαν να μην έχει γίνει τίποτα με τη Ρωσία, business as usual, είναι και αυτό ένα θέμα. Και τώρα θα δώσω το λόγο, λέει ο πρόεδρο, στην κυρία Γιατεμάκη για ένα λεπτό. Δεν βλέπω όμω να είναι εδώ η κυρία Γιατεμάκη, οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Πόσελ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Πούτιν είναι αντιδημοκρατικός και θα έπρεπε να είναι πολύ πιο οξύ ε, το ψηφισμά μας. Θέλω όμως ε, να τονίσω διάφορα θέματα τα οποία χρειάζονται για το μέλλον. Να υπάρχει ε, βελτίωση της δυνατότητας διαματηρίας της αντιπολιτεύσεως. Ελεύθερα μέσα ενημέρωσης γιατί μόνο έτσι θα διοργανωθούν ελεύθερε ελεύθερες εκλογές. Διαδικασία η οποία θα επιτρέψει να υπάρχει μία πολυμορφία και ε, να επαναληφθούν ε, οι ε, εκλογές της Δούμας πέρυσι διότι μόνο έτσι θα μπορέσει να υπάρχει δημοκρατία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στάκουλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ. Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πιστοί στις αξίες μας. Πρέπει σίγουρα να προχωρήσουν οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις στη Ρωσία και εμείς από την πλευρά μας πρέπει να φροντίσουμε η Ρωσία να, έχει κάποια στιγμή ελεύθερο ε, σύστημα ελεύθερων εκλογών. Εμείς πιστεύουμε ότι η Δούμα και ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν έχουν εκλεγεί νόμιμα με βάση τις δικές μας αρχές και αξίες και εκεί είναι και το πρόβλημα. Πρέπει η Ρωσία να μπει στην τροχιά της δημοκρατίας. Ε, ίσως πρέπει να πετύσουμε νέες εκλογές στη Ρωσία. Εδώ Πρέπει να επενθυμίσουμε ότι και το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, που στεγάζεται στο διπλανό κτίριο έχει ε, επίσης δηλώσει ότι θα πρέπει η Ρωσία να κάνει και αυτή τις προσπάθειές της και πολλά πρέπει να κάνει και ο πρόεδρος ε, Πούτιν. Ένα καλό στοιχείο και για τον ίδιο τον Πούτιν θα ήταν αν προκύρεται εκ νέου εκλογές. Δεν μπορεί να μείνει πια τόσα χρόνια στην εξουσία ο Πούτιν. Κυρία Ζαμπόρσκα τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ υπερψήφισα το ψήφισμα, αλλά θεωρώ ότι είναι επαρκέ. Περιγράφει τις ελλείψεις και τις παρατυπίες κατά την προετοιμασία και την διεξαγωγή των εκλογών, αλλά είμαι πεπισμένη ότι αυτές οι εκλογές ε, ε, ήταν οθευμένες. Εγώ έχω μεγαλώσει κομμουνιστική δημοκρατία και ξέρω τι σημαίνει να έχει κάποιο εκλογικό αποτέλεσμα περίπου 100%. Αντίστοιχα αποτελέσματα είχαμε σε αρκετέ περιοχέ στη Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι παγκόσμιος παίκτη μόνο όταν δεν επιτρέπει να την εκβιάζουν κατά αυτόν τον τρόπο. Εξαρτώμεθα μένα από τη Ρωσία για την ενέργειά μας και τις πρώτες ύλε, αλλά η Ρωσία ε, εξαρτάται και από εμά για τα δισεκατομμύρια που τους πληρώνουμε για τις πρώτες ύλε και την ενέργεια. Θα πρέπει λοιπόν ε, να τεθούν όροι και αν ο Πούτιν ε, θα ε, καταπιέζει ε, ειρηνικού διαδηλωτέ, θα πρέπει όπω και στην περίπτωση τη Λευκορωσία να λάβουμε μέτρα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Λαντσπέργη τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπερψήφισα κι εγώ το θέμα της Ρωσίας παρά το γεγονός ότι υπήρξε μεγάλη ε, διαφθορά στις εκλογές της 4ης Μαρτίου για την εκλογή του Πρόεδρου στη Ρωσία. Θα ήθελα εδώ να πω ότι τουλάχιστον μία τροπολογία η οποία κατατήθηκε η Α1 στο πρώτο τμήμα και ήταν πολύ σημαντική διαδικασία, αλλά δυστυχώς δεν υπερψηφίθηκε. Θα πρέπει, λέμε, να ληφθεί ε, σοβαρά υπόψη το γεγονόν ότι η διαδικασία επιλογής ενός Προέδρου ε, δεν μπορεί, εάν δεν γίνει υπό όρους, να είναι μια ανταγωνιστική και τίμια επιλογή. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στο ψήφισμα για το Καζακστάν. Ο κύριος Καμίνσκι. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, από γεωπολιτική σκοπιά, το Καζακστάν είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο λόγω της γεωγραφικής του θέσης, αλλά και για την ευρω... ευρύτερη ευρασιατική περιοχή. Το Καζακστάν μέχρι τούδε ήταν μια χώρα η οποία κατάφερε να αποφύγει τις εθνοτικές και θρησκευτικές συγκρούσεις που είναι πάρα πολύ συχνές σε άλλα μέρη του κόσμου. Ε, και το γεγονό ότι υπάρχει ανεξιθρησκεία στη χώρα ε, έπρεπε να μα κάνει να την εκτιμούμε ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό ακριβώ ε, ανησυχήσαμε ιδιαίτερα για τόσα συνέβησαν το περασμένο Δεκέμβριο. Είχαμε θανάτου ε, θανάτους σε διαδηλώσει απεργών και αυτό μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό δηλώνω ικανοποιημένος που οι αρχές του Καζακστάν όπως φαίνεται από τις πληροφορίες, έκαναν μία απόπειρα να τιμωρήσουν ε, όσους ήταν ένοχοι για τα όσα συνέβησαν και να τους δικάσουν. Εμείς θα πρέπει να αποστείλουμε το μήνυμα ότι η δημοκρατία είναι για όλους. Κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου και επομένως οι ένοχοι θα πρέπει να περνούν από δίκη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάναν. Δεν τον βλέπω όμως στην αίθουσα. Ένα λεπτό λοιπόν για τον κύριο Μέρφυ. Ε, Κύριε Πρόεδρε, η ομάδα μου, η Γκουε, προτείνει κάποιε τροπολογίε για να είναι πιο ισχυρό αυτό το ψήφισμα. Καταδικάζουμε τη νομή σφαγή που, διαπράττουν, που διέπραξαν μάλλον το Δεκέμβριο στο Πακιστάν οι αρχέ. Υπάρχει διωγμό τη αντιπολίτευση, υπάρχει παρενόχληση ε, των μέσων μέσων ανεξάρτητων δημοσιογράφων. Υποστηρίζω και την απεργία των εργαζόμενων ε, στον τομέα του πετρελαϊκού γιατί είναι τα αιτήματά τους ε, δίκαια και όλων των εργαζομένων δημοσιογράφων και αντιφρονούντων ε, τα δικαιώματα τα υποστηρίζω. Παρά την καταστολή εκφράζονται. Και τελικά πρέπει να πω ότι απήχα στην ψηφοφορία της εκθέσεως γιατί ναι μεν θέτει τα σωστά ερωτήματα και τις ανησυχίες για την ανησυχητική επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τελικά κάνει ε, τη χάρη στο καθεστώς του Καζακστάν ε, να γλυκένει λίγο, να χρυσώνει λίγο το χάπι, ενώ επιδεινώνει την κατάσταση να λέει ότι ναι, έχουν κάνει βήματα, πρόοδο κτλ. κτλ. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Όγγελαντ, για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος για το Καζακστάν. Χθες στην αίθουσα αυτή έγινε μια συζήτηση εντελεχέστατη για τα γεγονότα του Δεκεμβρίου στο Καζακστάν. Κανείς δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτά τα γεγονότα και όποιοι ήταν ένοχοι για τους ανθρώπους που πέρασαν τη ζωή τους πρέπει να παραπευτούν στη δικαιοσύνη. Το Καζακστάν βέβαια είναι μια σημαντική χώρα με πολύ σημαντικού πόρου, ε, με μεγάλη ισχύ. Άρα είναι προ το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί με τη χώρα αυτή. Βέβαια, προπόθεση για τη συνεργασία με το Καζακστάν πρέπει να είναι ο εκδημοκρατισμό του, του Καζακστάν. Ο πρόεδρο Νασαρπάκηφ έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να οδηγήσει τη χώρα του και το λαό του σε ένα καλύτερο μέλλον προς ε, τις δημοκρατικές αρχές. Κύριος ε, Τάνο, δεν πρέπει να υποτιμηθεί η κατάσταση. Έχουμε πολύ καλή σχέση με το Πακιστάν. Πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μα, ιδίω στον τομέα του διαλόγου για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το εμπόριο και την καταπολέμηση τη δημοκρατία, του εγκρανωμένου εγκλήματο και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Στηρίζουμε την έκκληση να καταβάλουν οι, αρχές του Καζακστάν κάθε προσπάθεια να διερευνήσουν ε, τις ε, πυροβολισμούς που έπεσαν κατά των εργαζομένων στο του πετρελαϊκού το Δεκέμβριο. Η ΟΑΣΕ έχει κάνει επίση συστάσει, οποίε υποστηρίζουμε. Θα πρέπει οι πυροβολισμοί από την αστυνομία να ερευνηθούν. Νομίζουμε ότι μεροληπτεί το ψήφισμα όμως ε, και μέχρι ότου είναι γνωστά όλα τα πραγματικά στοιχεία και περιστατικά, προτιμήσαμε εμεί να απέχουμε. Παραδόξω όπω και η Γκουε, αλλά τέλο πάντων οι λόγοι μα ήταν τελώ διαφορετικοί. Ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα στην κατάσταση στην Ιγυρία. Ο κύριος Στάτλερ έχει πρώτος το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι είναι μόνο ένα από τα προβλήματα που πρέπει να αναγνωρίσουμε διότι στις μουσουλμανικές χώρες υπάρχουν πολλές και μαζικές επιθέσεις κατά των χριστιανών και των κοπτών το ίδιο και στη Συρία και η κατάσταση έχει χειροτερέψει τελευταία και στο Ιράκ και στη Σαουδική Αραβία και οι χριστιανοί ε, είναι πλέον έχουν συρρυκνωθεί σε μία ε, ελάχιστη μειοψηφία και έχω γνωρίσει και πρόσφυγες στην Αυστρία. Υπάρχει λοιπόν θρησκευτική διαμάχη η οποία πλήττει τα αδέρφια μας εν Χριστώ και πρέπει να τους προσπαθήσουμε να τους υπερασπιστούμε. Ευχαριστώ πολύ κατά τη διάρκεια της επεξήγησης ψήφων ε, προς ενημέρωσή σας δεν προβλέπεται να χρησιμοποιείται η μπλε κάρτα. Ο κύριος Καμίνσκι τώρα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι χριστιανοί σήμερα ανά τον κόσμο είναι μια θρησκευτική ομάδα που αποτελεί αντικείμενο δίωξη και μάλιστα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό συμβαίνει δυστυχώ σε όλε τι υπέρου και όπω διαπιστώνουμε και στην Ιγυρία. Οι χριστιανοί λοιπόν και πολλοί από τους παρισταμένους νιώθουν αλληλεγγύη προς τα αδελφούς μας ε, στην Ιγυρία. Δεν μπορεί στον 21ο αιώνα να δεχόμαστε αυτά τα φαινόμενα. Αυτοί που λένε αγαπάτε αλλήλους, ε, οι χριστιανοί βρίσκονται να δολοφονούνται και να τους στερούνται τα δικαιώματά τους. Και θα πρέπει να πω ότι υποστηρίζουμε τους χριστιανούς αδελφούς μας στην Ιγυρία και με τις πράξεις μας και με τις προσευχές μας. Ο κύριος Μέρφη τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Μαζί με το αδελφό μου κόμμα στην Ιγυρία, το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κίνημα, ε, δικάζω τη βία του Μπόκα Χαράν. Αυτό το κίνημα δεν έχει να προσφέρει τίποτα στους εργαζομένους της Νιγηρίας, πέρα από θρησκευτικές και εθνοτικές ε, ε, περιπτώσεις βίας, βία μεταξύ ε, στρατιωτικών δυνάμεων και θα ε, δούμε και διεφθαρμένους πολιτικούς. η βία ε, βρίσκεται σε μαζικά κινήματα και θα πρέπει να ενοποιηθούν οι φτωχοί και οι εργαζόμενοι ενάντια όλων αυτών των οργανωμένων, ε, των πλουσίων και των μεγάλων επιχειρήσεων που κλέβουν όλο το ε, πλούτο της Νιγηρίας. Το 1% του πληθυσμού καταλυστεύει το 90% του πληθυσμού και τον αφήνει να ζει κάτω από το όριο της πτώχειας. Θα πρέπει λοιπόν ε, ε, να λάβουμε υπόψη μας τις διαδηλώσεις, οι οποίες δεν ήταν απλώς μια διαδήλωση απεργών, ήταν ε, έτοιμα για να σταματήσει η κατάσταση και να αλλάξει το καθεστώς. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουν αυτές οι διαιρέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πόσελτ είναι ο τελευταίος ομιλητής για το συγκεκριμένο ψήφισμα σε, στη μεγαλύτερη χώρα α, παραγωγής πετρελαίου στον κόσμο ο, καταδιώκονται οι χριστιανοί βία και αυτό το απέχει αποδείξει και η καθολική ε, εκκλησία και όλοι και αν δεν διακηρύξουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση ότι προσπίζουμε τους χριστιανούς αλλά είμαστε υπέρ του διαλόγου και υπέρ της θρησκευτική ελευθερίας αλλά αν εμείς δεν ενδιαφερθούμε για τους χριστιανούς ποιος θα το πράξει οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ανοίξει αυτό το κεφάλαιο θα ήθελα ακόμη κάτι πιο σαφές προς αυτή την κατεύθυνση εκ μέρους των υπευθύνων ευχαριστώ το τελευταίο σημείο είναι η επεξηγήση ψήφου για το Παγκόσμιο Φόρουμ για το νερό. Ο πρώτος ομιλητής είναι η κυρία Μιράντα. Δεν είναι στην αίθουσα, επομένως ε, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Στάτλερ. Herr Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε μία πολύ καλή και είχαμε μία πολύ καλή συζήτηση σχετικά με το έκτο φόρουμ για το νερό ε, και νομίζω ότι η ανακοίνωση της της ε, ε, Επιτρόπου ήταν πολύ καλή ότι ε, θα πρέπει να υπενθυμίσει σε ορισμένες χώρες ότι στερούν διότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια να εστερνιστεί ότι πρέπει να εξοικονομεί νερό και θα πρέπει να σκεφτούμε εάν στο μέλλον δεν πρέπει να έχουμε χωριστές κυκλοφορίες νερού δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική, ε, διαφορετική παροχή ε, για το πόσιμο είδωρ και ε, για το πόσιμο νερό δεν είναι, δεν είναι δυνατόν να πρέπει οι άνθρωποι να πίνουν το βιομηχανικό νερό σε ορισμένες περιοχές περιοχές. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καμίνσκι τώρα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Από 12 έως 15 Μαρτίου συνεδριάζουμε στο Στρασβούργο, ενώ στη Μασαλία ταυτόχρονα έχουμε το έκτο Παγκόσμιο Φόρουμ για το νερό. Συζητούνται ζητήματα ύψης της σημασίας για ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων του πλανήτη μας. Υπάρχουν περιοχές στην Αφρική όπου η πρόσβαση στο νερό παρεμποδίζεται, είναι ανύπαρκτη. Εξού και στηρίζω τη δήλωση ότι η πρόσβαση στο νερό είναι ένα από τα σημαντικότερα θεμελιώδη δικαιώματα, διότι το νερό είναι ζωή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ καλά κάνουν και δεσμεύονται για το θέμα αυτό. Επευκαιρία λοιπόν του Παγκόσμιου Φόρουμ για το νερό ελπίζω να είναι πάρα πολύ επικοδομητικές οι συνεδριάσεις και αποφάσει που θα λάβει. Πρόεδρος, θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μπασέσκου για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος διότι η βελτίωση τη πρόσβαση στο νερό βελτιώνει και το επίπεδο διαβίωση. Η αποτελεσματική διαχείριση του νερού είναι πολύ σημαντική, ιδίω ε, για τη μείωση της φτώχειας. Και πιστεύω ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην όλη συζήτηση για την εκρίζωση της φτώχειας. Πρέπει να προστατευθούν ε, οι πόροι, τα αποθέματα νερού. Και αυτό πρέπει να μπει και στην ε, ημερήσια διάταξη της Συνόδου Ρίο 20 στηρίζω την ιδέα για τη δημιουργία παγκόσμιων ε, σχεδίων διαχείρισης του νερού. Ταυτόχρονα βέβαια είναι απαραίτητο να επαναξιολογήσουμε και την χρηματοδότηση που θα πρέπει να είναι επαρκής γιατί πρέπει να μπορεί ο κόσμος να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Η ποιότητα του νερού για τη Ρουμανία είναι προτεραιότητα. Πολύ σημαντικό θέμα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του περιβαλλοντικού κεκτημένου. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Πόσελτ. Κύριε Πρόεδρε, την προηγούμενη εβδομάδα στη Ρώμη μπόρεσα να μελετήσω πόσο η ε, ΦΑΟ προετοιμάστηκε έντονα για αυτό το φόρουμ του νερού και πρόκειται για ένα βασικό θέμα για την ανθρωπότητα γι' αυτό και χαιρετίζω το ψήφισμα αυτό αλλά νομίζω ότι πρέπει να απασχοληθούμε πολύ πιο έντονα διότι το νερό δεν είναι μόνο πηγή ζωής αλλά και θανάτου όταν η στενότης και ανεπάρκεια του νερού οδηγεί σε διαμάχες και σε πολέμους και όπως είπε και η συνάδελφος Μπασέσκου χρειαζόμαστε μία διαχείριση του νερού μία και η ιδιωτικοποίηση των ε, υδατίνων πόρων πρέπει να έχει όρια. Είναι ένα αγαθό που ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα, γι' αυτό και υπερψήφισμα τη σχετική τροπολογία, γι' αυτό και δεν πρέπει να γίνει αντικείμενο καταπίεση σε αυτό το αγαθό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. τελευταίο ομιλητή είναι ο κύριος Τάνοκ. Η ομάδα μου είναι υπέρ του ψηφίσματος για το, το Παγκόσμιο Φόρουμ για το νερό. Σχεδόν ο μισός από τον ε, πληθυσμό των αναπτυσσόμενων χωρών δεν έχει πρόσβαση σε καθαρό νερό. 800 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν νερό το οποίο δεν ε, είναι ασφαλές ε, και παρά το γεγονός ότι η δημόσια υγεία και η περιβαλλοντική προστασία αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες για τη διαχείριση των υδάτων, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι αναγνωρίζεται και ο ρόλος της πρόσβασης σε καθαρό νερό και το πώς διασφαλίζει την ειρήνη και την συμφιλίωση σε περιοχές σύραξης και επίσης ε, μας ενδιαφέρει και η επιβεβαίωση διεθνών συμβάσεων ε, για το γεγονός ότι θα πρέπει να ε, υπάρχει κατάλληλη κατανομή του νερού και να μην υπάρχουν εθνικά σύνορα για το θέμα αυτό. Είναι μια βασική πολιτική πρόταση για όλες τις πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Περατώθηκε ο κατάλογος των ομιλητών. Διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 3.